Δεν έχουμε σημείο 2. ανακοινώσει του Προέδρου. Πριν μπούμε στην κανονική ημερήσια διάταξη, ήθελα λίγο να σας πω για τις εκλογές, μάλλον να μας πούνε για τις εκλογές στην Αλβανία. Ακούμε από τον ΟΑΣΕ διάφορες ειδήσει που δείχνουν ότι υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα στις εκλογές. Ε, στην προεκλογική εκστρατεία, στην εκλογική αναμέτρηση και σε άλλα τεινά. Και θα ήθελα να ακούσουμε πώς έχουν εκεί εξελίξει, γιατί είναι σημαντική η χώρα. Ε, αφού έχουμε διαπραγματεύσεις προενταξιακές και ο κύριος Κούκαν και ο κύριος Φλέκενστάιν ήταν εκπρόσωποι μας εκεί ε, που παρακολούθησαν τη διαδικασία προσέγγισης των κομμάτων στην Αλβανία και ήθελαν να το φροντίσουν και να το κοιτάξουν αυτό το θέμα. Και πριν τις εκλογές ε, το έπραξαν με επιτυχία, αλλά έχω την αίσθηση ότι η ίδια η εκλογική αναμέτρηση, η διαδικασία των εκλογών πήρε άλλη κατεύθυνση. Και έτσι πολιτικά ήταν αρκετά τεταμένα τα πράγματα. Βλέπω λοιπόν ότι ο ΑΣΕ για τα θέματα της ελευθεροτυπίας ε, λέει πολύ σκληρά λόγια για τα όσα έγιναν εκεί. Μιλάνε εδώ για εξαγορά ψήφων και νοθεία στις εκλογές. είναι ε, νοθεία με τα ψηφοδέλτια, με διάφορα δείπνα και ε, με μονομερείς επεμβάσεις της ε, διοίκησης, με πίεση που ασκήθηκε σε κρατικούς υπαλλήλους. δηλαδή για να τους συνετίσουν και να τους συμμορφώσουν πώς θα ψηφίσουν, χρησιμοποιήθηκαν δημόσιες υπηρεσίες για κομματικές σκοπιμότητες και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Εφορευτική Επιτροπή και τη Δεξαγωγή των Εκλογών. Υπήρξαν δυσκολίες λοιπόν, απειλές, απειλές κατά τη ζωής ε, ε, και σωματικές βλάβες σε 39 περιπτώσεις, σε 43 νοθείες και τα λοιπά, 32 άλλες περιπτώσεις, εκλογικά τμήματα. Ε, οπότε το πρώτο που έχει νόημα να το συζητήσουμε. Παρόν δεν ήμουν και δεν έχω άποψη, ούτε μπορώ να κρίνω τι συνέβη, αλλά ο κύριος Φλέκενστάιν κάτι λέει εκτός μικροφώνου. Πάντως θα ήταν πολύ καλό εδώ στην Επιτροπή μας να το συζητήσουμε και ενδεχομένως να δώσουμε το λόγο στους κύριου Κούκαν και Φλέκενστάιν να μας δώσουν τη δική τους εκτίμηση. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να ασχοληθούμε περαιτέρω με αυτό το θέμα. Ε, Ντουάρτε, έχεις το λόγο. Παίρνει το λόγο ο κύριος Φλέκενστάιν. Δεν άξιος που είπα, Έντουαρτ. Να, δεν με νοιάζει κιόλα. ευχαριστώ. Δύο λόγια για την ε, προετοιμασία των εκλογών στην Αλβανία βρίσκεται σε μια δύσκολη πολιτική περίοδο και εντάσεις η χώρα. Απέχουν εδώ και αρκετούς μήνες οι, τα μέλη της αντιπολίτευσης από την κοινοβουλευτικές εργασίες. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, μαζί με τον κύριο Φλέκινστάιν επισκεφθήκαμε την Αλβανία λίγο πριν τα Χριστούγεννα το Δεκέμβριο και έτσι μπορέσαμε να, να συμβάλλουμε στην επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο πολιτικών κομμάτων που παρουσιάστηκε πριν του Κοινοβουλίου της Αλβανίας και εγκρίθηκε ομόφωνα. Υπήρξαν τοπικές εκλογές με υπόβαθρο τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που μειώνει τον αριθμό των περιφερειών σε 61 σε σχέση με τη σημασία της εκλογικής αυτής αναμέτρησης για την χώρα. Θεωρήθηκε ως μία δοκιμή της ε, δημοκρατικής ολοκλήρωσης στην Αλβανία, χώρα υποψήφια που περιμένει να τη δοθεί η ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Άρα οι εκλογές αυτέ θα είναι πολύ σημαντικέ και είναι πολύ σημαντικέ για το μέλλον και την πρόοδο στην υπόθεση αυτή της Αλβανίας. Είχα επαφές με εκπροσώπους του διεθνή παράγοντα της ΟΑΣΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέσβυρα, Λαχούτιν, Αμερικανό πρέσβη στην Αλβανία, επίσης είδα. Ε, διάβασα τις προκαταρκτικές ε, εκθέσεις του ΟΣΕ. που σημειώνουν ότι υπάρχουν πολλές παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία και σε αυτά που αναφέρεις και εσύ Ελμαρ έγινε λόγος όμως και για πιο θετική διαδικασία την ημέρα των εκλογών, πιο θετικά δηλαδή, πιο θετική εικόνα την ημέρα των εκλογών, χωρίς σοβαρά προβλήματα κατά τη διεξαγωγή τους. Ε, θετικό μήνυμα επίσης ήταν το ότι εν γέννη τα πολιτικά κόμματα δέχθηκαν τις, ε, το αποτέλεσμα των εκλογών, ε, ο ιτημένος ε, συνεχάρη τον νικητή των εκλογών. Πάντως θα έλεγα ότι θα πρέπει κατά ψηφθαντά να συνεχιστεί η συζήτηση όταν θα έχουμε από τους διεθνείς φορείς τις τελικές εκθέσεις, εκείνους δηλαδή που είναι επιφορτισμένοι με την παρατήρηση των εκλογών. Πάντως εγώ μπορώ να σημειώσω τα εξής. Την αποποινικοποίηση τμήμα της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί και κατά την διάρκεια της παρουσίας του κυρίου Φλέκενστάιν και μου στη χώρα, δηλαδή την αποφυγή ε, χάρη νέα νομοθεσίας που έχει εισαχθεί στη, τη συμπερίληψη σε εκλογικές λίστες ανθρώπων που έχουν ε, καταδικαστεί για ποινικά δικήματα. Αυτό δεν επετεύχθη όπως θα έπρεπε εγκαίρως, στις επόμενες εκλογές θα το δούμε. Και επίσης η εξαγορά ψήφων για την οποία έγιναν αρκετές καταγγελίες και πρέπει να, να ε, διαρευνηθεί. Βέβαια αυτή η εξαγορά ψήφων ε, είναι δύσκολο να αποκαλυφθεί γιατί όποιος έχει δεχθεί να πληρωθεί για την ψήφο του κινδυνεύει να κατηγορηθεί και αυτός για ποινικό αδίκημα. Και έτσι δεν τολμάει κανείς να μιλήσει στην ε, αστυνομία. Αυτό θα ήταν μια σοβαρή παραβίαση. Η πολιτικοποίηση των κρατικών θεσμών και άλλα ζητήματα που αναφέρατε και εσείς επίσης έχουν τραβήξει την προσοχή μας οι εργασίες της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν φάνηκε να διεξήχθησαν κατά τρόπο απρόσκοπτο πάντοτε. Και εγώ θα έλεγα, Έλμαρ, πριν καταλήξουμε σε τελικά συμπεράσματα, να περιμένουμε να δούμε τις εκθέσεις της ΟΝΤΙΡ και της ε, ΟΔΟΑΣΕ για να δούμε το θέμα αυτό κατά τρόπο πλήρη και διεξοδικό, καθώς έχουν τεράστια σημασία για τις εξελίξεις της χώρας, στη χώρα αυτές οι εκλογές. Ευχαριστώ. Äh, Θα ήθελα να προσθέσω πολύ λίγα γιατί συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε ο κύριος Κούκαν. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι λέει ο, Γενικά, ήταν ε, κανονική η διεξαγωγή των εκλογών. Η δική μας αποστολή λέει ότι ήταν η καλύτερη από όλες τις προηγούμενες ε, εκλογική αναμέτρηση. Και οι πρεσβείες, η Ιταλική ας πούμε λέει ότι ήταν μια καλή μέρα για την Αλβανία, αλλά δεν θα πρέπει να γελιόμαστε. Αυτά που λέει εδώ ότι ε, συνέβησαν προφανώς και θα πρέπει να περιμένουμε ε, την τελική έκθεση για να ε, δούμε τι θα κάνει και η κυβέρνηση, γιατί περιμένουμε βελτιώσεις. Και αν χρειαστεί και επανάληψη των εκλογών, ε, δεν ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το αξιολογήσω, αλλά θα περιμένουμε. δύο πράγματα θεωρώ προβληματικά. Ένας πρόεδρος κόμματος έρχεται στη Βρυξέλλη στην πολιτική του παράταξη και λέει δεν αναγνωρίζω ε, το αποτέλεσμα, το εκλογικό. Γενικά, συλλήβδιν, αυτό είναι πολύ εύκολο. Να δούμε, ε, σε 61 περιφέρειες έγιναν εκλογές, ήταν τόσο μεγάλες και πολλές οι ατασταλίες κοινοθείες. Λοιπόν, εάν ναι, θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε αυτό. Ο Επίτροπος Χάν ήταν πολύ μετριοπαθής στις δηλώσεις του Είπε ότι περιμένει το τελικό αποτέλεσμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφανθεί με τη σειρά τη. Και εγώ θα ήλπιζα να είχαν αντιδράσει όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κανεί άλλο το λόγο. Ωραία. Θα ήθελα να ακούσουμε... Μάλλον το πω να προσκαλέσουμε τον εκπρόσωπο, ή τον εισηγητή του ΟΝΤΙΡ σε δύο μήνες ας πούμε που είναι το Γραφείο για τους Δημοκρατισμικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΑΣΕ και να καλέσουμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Τύρανα για διαβουλεύση, γιατί ακούω ότι έχει άποψη και ισχυρή ότι ας πούμε εκδηλώθηκε, πήγε και σε κομματικές ε, εκδηλώσεις από ό,τι άκουσα. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να αποδειχθεί ενδεχομένω ε, εσφαλμένη είδηση, λάθος. Λοιπόν, συμφωνείτε. Καλώς. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι... Gipfel ο συνάδελφος Ντανζόν αποσιάζει να μας πει για τη Σύνοδο κορυφή. που κανονικά έπρεπε να ασχοληθεί με την άμυνα και την ασφάλεια την περασμένη Πέμπτη του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο. κατά κύριο λόγο και ουσιαστικά επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2013 και τώρα θα πρέπει κανείς να αξιώσει να εφαρμοστούν και με τη συζήτηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με την κυρία Μογκερίνη αυτό θα αφορά πλέον τον Ιούνιο του 2016 για τη στρατηγική που θα καταδεθεί γενικότερα, τη συνολική μας στρατηγική. Ε, στην συνεδρίαση των συντονιστών προηγουμένως αποφασίσαμε να γίνει μια έκθεση σχετικά, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό και ε, ε, καλό θα ήταν εγκαίρως εμείς να παρέμβουμε σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στενότερη συνεργασία για την αμυντική συνεργασία ιδιαίτερα και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα πρέπει να μας απασχολήσει συνδυασμένα η συζήτηση στην έρευνα και την τεχνολογία σε υβριδικές απειλές, σε θέματα συνεργασίας αμυντικής βιομηχανίας είναι σαφή τα πράγματα. Βέβαια δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες, δεν έγινε ευρία συζήτηση, δεν επεκτάθηκαν σε αυτό. Είναι γεγονός γιατί τον Οκτώβριο το που μας πέρασε κυριάρχησαν άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη, ε, όπως το Brexit π.χ. Όπως είχαμε φράσει φόβου στην περασμένη Τρίτη, ε, δόθηκε μια μικρή εντολή που είχαμε αποφασίσει και εμείς στις εκθέσεις μας για την εξάντληση των δυνατοτήτων που παρέχει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ιδιαίτερα η Μεγάλη Βρετανία απέριψε την παραμικρή νήξη σε αυτό το θέμα. Και επειδή το Ευρωπαϊκό αυτό Συμβούλιο πρέπει πάντα να αποφασίζει ομόφωνα, έχουν τα πράγματα όσοι έχουν. Αν δεν είμαστε πια καν σε θέση να συζητάμε τέτοια θέματα, για αρμοδιότητες των συνθηκών, να τα κατονομάζουμε για να διερευνούμε τη δυνατότητα εφαρμογής τους, ε, ε, λόγω και των ε, παρόντων προβλημάτων και προκλήσεων στην πολιτική ασφαλείας, τότε έχουμε μπλέξει για τη μεταξέλιξη. Δεν υπάρχει κανένα πεδίο που να έχουμε υποστήριξη ε, του λαού σε όλα τα κράτη-μέλη ε, όσο για την ασφάλεια. Ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η Ευρώπη. Συμφωνούν οι πολίτες αυτό. Και ήταν αυτό ένα καλό μήνυμα προς Ανατολάς. Πώς το βλέπει η Ανατολή αυτό. Αυτή η εμπλοκή δηλαδή ήταν ενθαρρυντική για αυτούς. Και λόγω τη ομοφωνία στο Συμβούλιο δεν πρόκειται να προχωρήσει. Και υπάρχουν δικέ μας εκθέσεις που έχουμε αποφασίσει και στην Επιτροπή μας κατά πλειοψηφία και στην Αλομέλεια και ε, θα πρέπει να τις προωθήσουμε. Γιατί εδώ παίρνουμε αποφάσεις με μεγάλη πλειοψηφία τις οποίες κάποιοι αγνοούν. Μιλούσαμε για ανάθεση εντολή στην ύπατη εκπρόσωπο να διερευνήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την εξάντληση των δυνατοτήτων που απορρέουν από τις συνήθειες της Αβώνας και τίποτα παραπάνω. Δεν αναφέρουν καν τη λέξη των πέντε γραμμάτων πέσκο. Δηλαδή και αυτό για να γίνει συμβιβασμό πρέπει να παρακαμφθεί. Μα ε, δεδηλωμένο στόχος ήταν να προχωρήσει η ε, συμμαχία των προθήμων και να υπάρχει μια νόμιμη μόνιμη ε, επιτροπή και συνεργασία και αυτό ήταν κόλαφος για την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και για τα όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Στη Ρίγα ήμουν χτες παρόν σε μια συζήτηση μεταξύ ευρωβουλευτών και ε, Αμερικανών γερουσιαστών Ξέρετε ότι κάθε εξάμεινο έχουμε συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν το Κογκρέσο και εμείς ζητούμε από τους Αμερικανούς να φροντίσουν να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια, περισσότερη ασφάλεια στην Ανατολική Ευρώπη και πού είναι η διαστρωμένη συνεργασία και η συλλογική άμυνα. Μόνο με το ΝΑΤΟ υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οπότε τίθενται ερωτήματα και εσείς τι κάνετε. Και η απάντησή μας είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, δεν θα αποφύγουμε εμεί στενότερη συνεργασία και θα πρέπει να απευθύνουμε και αυτό το ερώτημα προς τις νέες χώρες, ανατολικά κράτη, που έχουν ιδιαίτερο συμφέρον και ενδιαφέρον, αλλά δεν αντιτάχθηκαν σε αυτή τη βρετανική πρόταση. Υπήρχε μία χώρα που ήθελε να μπει, αλλά μετά της είπαν ότι οι Βρετανοί έχουν δημοψήφισμα και υποχώρησε. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να έχει θετική έκβαση το Βρετανικό δημοψήφισμα. Γιατί εγώ εκτιμώ πάρα πολύ την παραμονή της, Ευρωπαϊ... της ε, Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορούμε να παραλύσουμε για δύο χρόνια τώρα να ε, ε αποκλειστεί οποιαδήποτε δυνατότητα μεταξέλιξης και συνεργασίας. Αυτά. Έχετε παρατηρήσεις από αυτό. Με εκπλήσει που δεν ζητεί κανείς το λόγο επ' αυτού. Παρακαλώ. Auch die EVP nicht. Το ΕΛΚ κανείς. Η κυρία που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Ε, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν θέλετε να μιλήσω γενικά ή μόνο για την άμυνα. Μισό λεπτό γιατί δεν ακούω τίποτα. Ε, έλεγα, Πρόεδρε, ε, χρειάστηκε να βγω γιατί είχα μια τηλεφωνική συνομιλία. Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Άμυνα. Αυτό ε, τώρα θα τα πω ή θέλετε να περιμένω. Τώρα, τώρα, τώρα. Θα τα πω στα Ολλανδικά γιατί είναι πιο εύκολα για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σύντομη ενημέρωση, Πρόεδρε. Και εγώ περίμενα αυτή η σύνοδο κορυφή να μπει στην ουσία των θεμάτων άμυνας και ασφάλειας. Αν κοιτάξετε το Δεκέμβριο του 2013 τι είπανε, είχε δημιουργηθεί η ελπίδα ότι ε, θα ε, προχωρήσουν, αλλά διαψεύστηκε αυτό από την πραγματικότητα. Εμείς από τους φιλελευθέρους θεωρούμε σιγά σιγά ότι άμυνα και ασφάλεια δεν βρίσκουν τη σημασία που θα τους άξιζε ε, στα μάτια του Συμβουλίου. Μετά από 1,5 χρόνο επιβεβαιώνουν, λέει, ε, αυτά που αποφάσισαν το 2013 και αναβάλουν την επόμενη απόφαση για το επόμενο Συμβούλιο Κορυφής. Το 2016 θα έχουμε μια συνολική στρατηγική, λέει, ε, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και πρέπει να σας πω ότι επιτέλους καιρός ήταν μετά από 13 χρόνια. Μπράβο μας, θα έχουμε ε, ενημέρωση και αναβάθμιση του σημείου μας Σολάνα. Πάλι καλά. Και πάλι ε, ε, αυτού θα πρέπει να οικοδομήσουμε τη στρατηγική μας. Ως ομάδα εμείς δεν περιμέναμε ε, τα αποτελέσματα του Συμβουλίου. Την περασμένη εβδομάδα καταθέσαμε ένα σχέδιο, ALDE, οδικό χάρτη, προς μια ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη άμυνα. Και κάνουμε αυτή την πρόταση μαζί με τους φιλελεύθερους υπουργούς αμήνης Τσεχίας και Ολλανδίας και της Φιλανδίας, ένα πρώην υπουργό, ε, είναι ρεαλιστικό το σχέδιο, είχε πολύ θετικό αντίκτυπο. Εμεί θέλουμε οπωσδήποτε να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό σκέλος του ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει να έχουμε και κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το δόγμα Σολάνα χρειάζεται ενημέρωση ε, για μια ενοποιημένη στρατιωτική δυνατότητα και με κάθε ειλικρίνεια να δούμε τα πράγματα ε, κατάματα. Αυτά που δαπανούν τα 28 κράτη-μέλη, αν τα συγκρίνουμε με τον προπολογισμό ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μου πείτε τα νούμερα είναι νούμερα, αλλά είναι και εύλογα. Αν το προσθέσετε λοιπόν, είναι 45% με αποτέλεσμα, του αμερικανικού προπολογισμού με αποτέλεσμα 15% των δυνατοτήτων των Αμερικανών. Οπότε τα λεφτά μας δεν πιάνουν τόπο. Χρειάζεται περισσότερο συνοισμός και εμείς οι φιλελεύθεροι θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα. Και τα αποτελέσματα της περασμένης εβδομάδας μας έδειξαν κατάφορα ότι θα πρέπει να δραστοποιηθούμε και όλα τα κόμματα εδώ στην Επιτροπή μας να ε, μελετήσουν παρακαλώ τον οδικό χάρτη Άλντε και να μας δώσουν ε, τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κάποια σχόλια. Στο όπως και όλοι οι άλλοι, απογοητευθήκαμε κάπως με το, από το γεγονός ότι το πλαίσιο της του τελευταίου Συμβουλίου ε, στην ουσία απομακρύνθηκε από τις προτεραιότητες ε, που είχαν οριστεί ως θέμα, κύριο θέμα της ε, διάσκεψης κορυφής, γιατί το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, το θέμα της Ελλάδας και ανακοίνωση του δημοψηφίσματος της Ελλάδας κάπως επισκίασαν τα πολυαναμενόμενα πορίσματα για την ΚΕΠΑ. Εγώ πιστεύω πως η υπόθεση της κοινής εξωτερικής, της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας δεν είναι κάτι όνειρα από τη θερινής νυχτός, είναι κάτι πιο ουσιαστικό και όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε ε, για την, ε, καθολική, τη νέα καθολική στρατηγική για την άμυνα και την ασφάλεια που θα βασιστεί σε τρεις εκθέσεις που είχαμε για την ΚΕΠΑ, την άμυνα και την άλλη για τη χρηματοδότηση της ΚΕΠΑ και νομίζω και ξέρω πως το ΕΛΚ θα το συζητήσουμε αλλά φαντάζομαι και οι άλλες ομάδες θα τα συζητήσουν εμείς θα το συζητήσουμε το φθινόπωρο και θέλουμε γρήγορα να υπάρξει κάποια αντίδραση, συγκέντρωση των πόρων γιατί οι απειλές είναι προφανείς και όπως είπατε η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ είναι ένα από τα θέματα κλειδί. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχουμε αρκετά σημεία, αρκετά πορίσματα, ε, η τελευταία φράση που λέει ότι θα το διατηρεί στην ημερήσια του διάταξη του Συμβούλιο μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπιστεί πιο ουσιαστικά και μεγαλύτερη αξιοπιστία. Γι' αυτό και πιστεύω πως όλες οι ομάδες θα πρέπει να διατηρήσουν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Βάσμαν ε, είπε ότι οι Αμερικανοί δαπανούν 35% ενώ οι Ρώσοι 65% δαπανούν για τους ίδιους ίδιους στόχους, αντίστοιχα. Αλλά αυτοί αγοράζουν τάγκς. Εμείς εκθέσεις αγοράζουμε. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν 182 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για την αμυνά τους. Πολύ περισσότερο από ότι η Ρωσία. Και διαθέτουμε και, 200, ε, και διπλάσιους στρατιώτες από την Αμερικανία. Υπάρχουν όμως αυτές οι συνεργατικές σχέσεις, ο συνδυασμός των δυνάμεων. που πρέπει να αναπτυχθεί, γιατί έχουμε μόνο 10% του αποτελέσματος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Σπαταλάμε τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου με πολύ ψηλό κόστος. Η διοίκηση λειτουργεί από μόνη της, δεν χρειάζεται να έχουμε τόσους πολλούς στρατιώτες και το πρόβλημα που έχουμε είναι σαφές. Αλλά βέβαια καταλαβαίνω και ότι οι συνάδελφοι δεν συγκινούνται τόσο πολύ. Γι' αυτό και θα κλείσω εδώ τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ θερμά. Και πάω στο επόμενο θέμα τη ημερησία τάξη. Αλλά θα ξαναπώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ξαναδούμε. Αν υπάρχουν ε, ζητήματα τα οποία μπορούμε χωρίς να έχουμε έγγραφο ε, να υποστηρίξουμε, να συζητούμε γιατί έχουν επικαιρότητα. Έχει κανένα νόημα να κάνουμε ανταλλαγές απόψεων έτσι. Χωρίς ουσία, διότι αυτό μειώνει και την ε, αξία της Επιτροπής μας. Από την άλλη να κάνουμε ε, εκθέσεις με 450 τροπολογίες και να θεωρούμε ότι αυτό είναι πολιτική, πάλι δεν είναι σοβαρό. εξωτερική πολιτική είναι και η δυνατότητα να τοποθετείται κανείς για τα επίκαιρα θέματα και όχι μόνο να λαμβάνει εκθέσεις ε, που ενδιαφέρουν μόνο φοιτητέ. Άλλη βάση Και βλέποντας ότι αυτό δεν προξενεί μεγάλες συγκινήσεις, προχωρώ στο θέμα των σχέσεων με την ε, Ρωσία. Λευκό. Λευκορωσία. Τι μου στάτε το λόγο κύριε Φόλμαν. Ναι πρόεδρε. Εγώ χειροκρότησα την πρότασή σας γιατί ανισχύεται και θεωρώ ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να δώσει περισσότερη προσοχή από ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα και έχετε την υποστήριξη της Άλντε πλήρη σε αυτή την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς περνάω λοιπόν στο σημείο 4 της ημέρας διάταξης. Η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου επισκέφθηκε τη Λευκορωσία με τον κύριο Στροπιέσκη. Πρώτη, ύστερα από πολλά χρόνια ήταν η επίσκεψη αυτή. Και είναι νομίζω χρήσιμο να ακούσουμε μία έκθεση για την επίσκεψη αυτή της αντιπροσωπείας, αν ήταν χρήσιμη, πώς διεξήχθησαν οι συνομιλίες και αν κάτι άλλαξε. Έχετε το λόγο αγαπητέ συνάδελφα. Σωτροσκή, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Και ξεκινώ λέγοντας ότι σας έχουμε αποστείλει ανακοινωθέν και διάταξη των εργασιών αυτής της επισκέψεως. Άρα πρέπει να γνωρίζετε εν γέννη ποια ήταν η βασική ιδέα και τα θέματα που είχαμε να συζητήσουμε, ε, τι συναντήσεις και πόσες είχαμε να κάνουμε με την ε, πλευρά της κυβέρνησης, πόσες με την αντιπολίτευση. Διεξήχθη με βάση το σχέδιό μας και χωρίς δυσκολίες ε, η επίσκεψη, χωρίς εκπλήξεις ούτε δυσάρεστες ούτε ευχάριστες. Ε, για μένα ήταν σκόπιμη και χρήσιμη η επίσκεψη. Το πιο σημαντικό ε, για μένα ήταν ότι μπορέσαμε επανειλημμένως να υπογραμμίσουμε την ανάγκη και σεβασμό των βασικών αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι σε αυτό είμαστε ασυμβίβαστοι ε, το ζήτημα δηλαδή των πολιτικών κρατουμένων, το ζήτημα του υπομνήματος για την θανατική ποινή, το ζήτημα των δυσκολιών προς τη λειτουργία του, της δημόσιας διοίκησης στη χώρα, αυτά προς την κυβερνητική πλευρά. Συνομιλήσαμε όμως και με την αντιπολίτευση, οικογένειες αντιφρονούντων, πολιτικών κρατουμένων, επιχειρήσεις ε, που δραστηριοποιούνται στη Λευκορωσία και εκπροσώπους πολιτικών ομάδων και οργανωμένων πολιτών που ε, είναι γνωστοί και γνωστές για τις δραστηριότητες τους στην Ευρώπη αλλά και ε, διεθνώς. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι η Λευκορωσία είναι διατεθειμένη να συνομιλήσει μαζί μας. Υπάρχουν θέματα όπως η δυνατότητα κυκλοφορίας χωρίς υποχρέωση θεώρηση διαβατηρίων, οθέτηση των προτύπων ε, και προδιαγραφών της Μπολόνια, ζητήματα υποτροφιών με το σύστημα του Εράσμους, αρνητική εμπειρία μπορώ να πω ότι ήταν αυτή των συνθήκων ε, κράτησης των ολίγων πολιτικών κρατουμένων της χώρας. Πρέπει να συνεχιστεί, αυτό το επισημάναμε εμείς στην ε, κυβερνητική πλευρά, πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και πρέπει να ζητούμε βελτίωση ε, της κατάστασης και στον τομέα αυτών. Ε, το φθινόπωρο να μένετε να δεξαχθούν προεδρικές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος και οι συνθήκες υπό τις οποίες θα διεξαχθούν αυτές οι εκλογές. Αυτά εν ολίγης, εκ μέρους αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, εκ των οποίων δύο είναι παρόντες, η κυρία Κανιέτε και ο κύριος Μανίτης, αλλά και τους λοιπούς συναδέλφους όλου, και όλους όσους συνέβαλαν, όσοι συνέβαλαν, ε, με υποστήριξαν πολύ κατά την παραμονή μας στο Μίνσκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος μιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιο από τους προβληματισμούς μου και τις σκέψεις μου. Ε, πρόκειται για τη δεύτερη μου φετινή επίσκεψη στη Λευκορωσία. Την πρώτη φορά πήγα ιδιωτικώς και πήγα στο Υπουργείο Εξωτερικών και ασχολήθηκα με τη θέση των πολιτικών κρατωμένων στη δεύτερη μάλλον φορά, σε σύγκριση με την πρώτη μου επίσκεψη θα πρέπει να σας πω ότι είχα την εντύπωση, αποκόμισα την εντύπωση ότι η κατάστασή τους έχει επιδεινωθεί. Διότι τρει εξ αυτών ε, πέρασαν από περαιτέρω δίκες και ο φυλακισμός τους έχει παραταθεί. Η φυλάκισή τους έχει παραταθεί. Ε, Πίσω από άλλες πηγές μάθαμε ότι ο πρόεδρος Λουκασένκο είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην Λευκορωσία. Πράγμα που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από μια θέση που είναι αρκετά δύναμη, ούτε από λίγους πολιτικούς κρατούμενους που βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα. Η εντύπωση που είχα λοιπόν ε, ε, από τις συζητήσεις με συναδέλφους είναι ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι κατά κάποιο τρόπο είναι όμοιροι σε αυτό το ε, λεπτό παιχνίδι που παίζει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία. Κρατώντας τους σε σκληρές συνθήκες, στέλνει ένα μήνυμα τον ε, πρόεδρο Πούτιν, τον εταίρο του στη Ρωσία, ότι κοίτα δεν άλλαξα, είμαι ο ίδιος. Ωστόσο πρόκειται για ανθρώπους, ανθρώπινα όντα, που έχουν ε, μετατραπεί σε πιόνια, στη σκακέρα, του Λουκασέγκο και του Πούτιν. Πράγμα το οποίο με λυπεί ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα μετά από τα όσα άκουσα στη συζήτηση με τις οικογένειες τους. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι η αντιπολίτευση φοβάται ότι από τη μια πλευρά θα μπορούσε να υπάρξει ένα είδος ε, μετατραπής της Λευκορωσίας σε ένα είδος Αφγανιστάν, ε, Αζερβαϊτζάν με συγχωρείτε, και ότι ε, στην αντιμετώπιση του Λουκασέγκο ε, με την αντιπολίτευση ή τους πολιτικούς κρατούμενους όλα αυτά θα επισκιαστούν από κοινά ρεαλιστικά συμφέροντα. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι πως εν γέννη η αίσθηση που επικρατεί στην Λευκορωσία είναι ότι είναι περήφανοι για την ε, ανεξαρτησία της ε, χώρας τους και θεωρούν τον Λουκασέγκο τον μόνο πολιτικό που είναι σε θέση να καταφέρει να διατηρήσει την ανεξαρτησία της Λευκορωσίας. Και τα αιτήματα που είδαμε από ε, αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν αυτά. Παρακαλούμε να μην επιτρέψετε τη Λευκορωσία να επισκιαστεί από, άλλες, από άλλα μάλλον ευρωπαϊκά προβλήματα στην ε, ευρύτερη ε, περιοχή μας. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. I speak Latvian. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω λετωνικά και θα ήθελα Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου. Ήμουν στο Μίνσκ τον ε, Δεκέμβριο ιδιωτικό και είχα την αίσθηση πως η Λευκορωσία είναι ένας εταίρος για τη χώρα μου και τις υπόλοιπε αυτές τις χώρες, ε, τις δικές μας χώρες, ε, εκτός που είναι και γείτονα χώρα. Αλλά βεβαίως είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τις σχέσεις με την χώρα αυτή, γιατί όταν ας πούμε μιλάς με κάποιον, με κάποιον, της οποίας είναι στη φυλακή. Εκείνη είχε ένα ατύχημα και μόλις που γλίτωσε, δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι το ατύχημα αυτό ήταν ε, τελείως τυχαίο. Και επίσης γιατί δεν μπορεί να συνοηθεί η αντιπολίτευση να προτείνει έναν μόνο υποψήφιο. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί και κόμμα καταρχήν. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη συγκυρία, δεν υπάρχει προοπτική να έχουμε έναν μόνο υποψήφιο από πλευράς της αντιπολίτευσης. Εν τω μεταξύ όμως συμφωνώ μαζί σας ότι ο πρόεδρος Ρουκασένκο είναι πολύ δημοφιλής, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο η Κεντρική Επιτροπή, η Φοριστική Επιτροπή όντως θεωρεί πως το πραγματικό αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο φάνηκε. Να δούμε δηλαδή σε ποιο βαθμό υπάρχει εκδημοκρατισμός. Υπήρξε αντίσταση στον πειρασμό να αυξήσουν το ποσοστό Είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις συνομιλίες με τη Λευκορωσία ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το να υπάρχει μια, να έρθει μάλλον μια επίσημη ε, αντιπροσωπεία εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο είναι κάτι που δεν έχει συμβεί εδώ και 12 χρόνια και Και τέλος, δεν μπορούμε να ε, ε, συζητήσουμε ο καθένας λέγοντας τη δική του γνώμη σε αυτά τα ζητήματα υπάρχει, όπου υπάρχει ε, συμφωνία μεταξύ μας. Να σας πω ότι επισκέφθηκα ένα εργαστήριο για, που ελέγχει την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό εξοπλίστηκε με χρήματα ευρωπαϊκά και οι επιστήμονες έχουν πολύ θετική άποψη για αυτού του είδους τη συνεργασία. Για να μην ξεχνάμε βέβαια και άλλα σημαντικά είδη συνεργασίας που ήταν επιτυχή, όπως ας πούμε η καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, η βελτίωση των ε, συνοριακών ελέγχων, η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο διάλογος λοιπόν και η συνέχιση αυτού μπορούν να είναι ε, θετικός, να οδηγήσει σε επιτυχίες και φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε ως πρώτη προτεραιότητα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Thank you, Chairman. <clears throat> Well, I do agree that we have to keep Κύριε Σαστρεβίτσιος, πρόεδρε, συμφωνώ ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε το διάλογο μεταξύ ημών και Λευκορωσίας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει και να οξοδρομούμε σε σχέση με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επουδενή. Φαντάζομαι ότι αυτές ισχύουν ακόμη. Άρα δεν υπάρχει αναγνώριση των λεγόμενων εκλογών στη Λευκορωσία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πολιτικά εγκλήματα που έχει διαπράξει το καθεστώς του Λουκασέγκο. Μην ξεχνάμε δε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ε, χειριστικό πολιτικό μεγάλου βεληνικούς και μάλιστα το πρώτο δεξί του χέρι, μια γυναίκα που είναι επικεφαλής της ε, ε, επικεφαλής της ομάδας που είναι υπεύθυνη για κάθε είδους παρατυπία κατά την εκλογική εκστρατεία, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για εκλογές για να είμαστε ειλικρινείς, πώς θα τις ονομάσουμε εκλογές αν δεν μπορεί κανείς να, να ε, καταθέσει τα στοιχεία για να ε, συμμετάσχει σε εκλογές πολιτικό κόμμα, αν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στις εκλογές και μετά τις εκλογές τους ή άλλους παραμένουν στη φυλακή οι υποψήφοι, όπως συνέβη με τις προεδρικές εκλογές. Τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα λοιπόν. Και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την ε, επαφή με την αντιπολίτευση όσο αδύναμη και αν είναι, όσο διαλυμένη και αν είναι λόγω της πολύ πιο σαφούς συμμετοχής και εμπλοκής του καθεστώς του Λουκασέγκο στα γεγονότα αυτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε, ε, δεν πρέπει να υπάρχει καμιά περίπτωση να νομοποιήσουμε το καθεστώς του Λουκασέγκο και βαδίζουμε πάνω σε πολύ ε, αβέβαιο έδαφος. Όταν ο ίδιος ο Λουκασέγκο ευθύνεται για την θανάτωση δύο ατόμων ε, που καταδικάστηκαν για λόγους τρομοκρατίας υποτίθεται πέρυσι, δύο νεαρούς που θεώρησε ότι μπορεί να αξιοποιήσει ως θύματα για να μπορέσει να προβληθεί ως ισχυρός ηγέτης. Θεώρησε ότι μπορεί να θυσιάσει ο Λουκασένκο για να προβληθεί ως ισχυρός ηγέτης. Και φρονώ ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να δεχθεί δεν θα έπρεπε να έχει δεχθεί ε, εκπροσώπους της κάτω βουλής. Συνέβη όμως αυτό. Ήταν τρεις παρόντες από την κάτω βουλή. Δεν μου αρέσουν αυτά εμένα. Και σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν είναι δυνατόν να συναντιόμαστε με ιδιορισμένους από τον Λουκασένκο. Λάθος μηνύματα στέλνουμε και στην αντιπολίτευση και στην κοινωνία των πολιτών. Τι χρειάζεται πριν από τις εκλογές του Λουκασένκο χρειάζεται να δοθούν οι αναγνωρίσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αβέβαιο έδαφος λοιπόν μπορεί μερικές φορές να οδηγεί σε κατολιστήσεις. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και μπορεί από το αβέβαιο έδαφος να βρεθούμε και σε πολύ βαθιά νερά. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πολωνικά για να τα πω καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε, στη σημερινή συζήτηση μιλάμε για τη Λευκορωσία σαν να ήταν η Βόρεια Αφρική, σαν να ήταν καμιά απικία. Την κοιτάμε υποτιμητικά και προσπαθούμε να επιβάλλουμε αντιευρωπαϊκές αξίες, αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ήμουν από τη Λευκορωσία θα έλεγα δεν συζητώ μαζί σας περιφρονώ τους ανθρώπους που κατήργησαν τη θανατική ποινή. Γιατί ε, αυτοί έχουν άλλες αξίες από τις δικές μας. Έχουν τα χέρια τους αιματοβαμμένα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άλλες αξίες στη ζωή. Οι δικές μας αξίες δεν είναι οικουμενικές και πανανθρώπινες. Θα πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι οθούμε τον Λουκασέγκο στην αγκαλιά της Μόσχας. Ας προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο σενάριο. Εμείς τους πρόχνουμε τώρα στην αγκαλιά της Ρωσίας. Και αυτή είναι η βασική πολιτική αλήθεια πίσω από την τρέχουσα κατάσταση. Αν εσείς αποκαλείτε τους αυτούς σας δημοκράτες, εγώ δημοκράτης δεν είμαι, πρέπει να καταλάβετε ότι αν 75% του λαού υποστηρίζει τον κύριο Λουκασέγκο, εσείς που είστε δημοκράτες θα πρέπει να το τιμήσετε αυτό, έτσι δεν είναι. Αυτά είχα να σα πω. Και σα ευχαριστώ. χωρί μικρόφωνο, πρόεδρο. Yes. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Kiedy Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μόνο να πω ότι η αντιπροσωπεία μας δεν ε, συνάντησε βουλευτές που εξελέγησαν που εξελέγησαν ε, στις τελευταίες εκλογές. Υπάρχει μια κάποια ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες ε, συναντήσεις στην ημερησία διάταξη. Ήρθαμε σε επαφές με τις αρχές αλλά και με όσους αντιπροσωπεύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οικογένειες πολιτικών κρατούμενων, την κοινωνία των πολιτών και άλλους οργανισμούς ή ενώσεις που αναδύονται και φαίνονται να είναι ανεξάρτητοι. Υπήρξαν καλύτερες συνεδριάσεις και χειρότερες ε, όπου οι αξίες μας ε, δεν είναι κοινέ ούτε με την Εθνική Εφορευτική Επιτροπή ούτε με το Υπουργείο. Αλλά και εκεί συνομιλάμε συνομιλούμε ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εισακουγόμαστε. Είναι σημαντικό να εξακολουθήσουμε να ζητάμε καλύτερη μεταχείριση των πολιτικών κρατούμενων μεταξύ άλλων ε, για τα οποία ποτέ δεν πρόκειται να κάνουμε επίσης να συμβιβαστούμε και να ερχόμαστε διαρκώς σε επαφή με, τις, ε, ε, με τον κόσμο ώστε ο κόσμος και όχι οι αρχές να είναι ευπεπισμένοι ότι μας ενδιαφέρει το μέλλον τους. Το θέμα λοιπόν της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιουνίου. Για να δούμε. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Τμπράφκα Σουίτσα να αναλάβει, να μας το παρουσιάσει ως συγχυτρία. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως βλέπετε, έχω εκπονήσει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια Αδριατικής Ιουνίου, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είχα αντίστοιχα μια γνωμοδότηση για το ίδιο θέμα. Ξέρουμε ότι πρόκειται για μια έκθεση προτάσεως εκθέσεως της Επιτροπής Ρέτζι των Περιφερειών, ε, Περιφερειακής Επιτροπής, με εισηγητή τον κύριο ε, Γιάκοβτζιτς. 70 εκατομμύρια πολίτες θα ωφεληθούν από κάθε δυνατό πλεονέκτημα που θα προσφέρει η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η βελτίωση του βιώσιμου τουρισμού και άλλες πτυχές αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Για μας τώρα, για την εξωτερική πολιτική, θα βοηθήσει ιδιαίτερα τα κράτη που είναι ενδεχομένως ή δυνάμη υποψήφια, ώστε να αναπτύξουν τις δυνατότητες συνεργασίας, με τα κράτη-μέλη και βέβαια θα βελτιώσει και την ενοποίηση, την ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών της Δυτικής Βαλκανικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η πρώτη ευκαιρία που μπορούν να έχουν τα κράτη όπως η Αλβανία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία, η Ζεγοβίνη να συνεργάζονται με την Κροατία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία που είναι μέλη της Ένωσης. Η 9η Μαΐου, όπως ξέρουμε, ήταν η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών, κατατέθηκαν 47. Τετάρτη 1η Ιουλίου γίνεται μια συνεδρίαση για να ε, συνομιλήσουμε και να ορίσουμε κοινέ τροπολογίε. Ε, συμβαστικές, ελπίζω με τους σκιώδες συγκητές. Είμαι βέβαια ότι έχετε όλοι αναγνώσει την ε, γνωμοδότηση, ξέρετε ότι υπάρχει περιορισμός προς τον αριθμό των λέξεων. Ξέρετε ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν γενικά για την εκπόνηση γνωμοδοτήσεων, δηλαδή δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε όλα τα θέματα που θα μας ενδιαφέραν. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε χάρη στην κατάθεση τροπολογιών να την συμπληρώσουμε. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ε, το θέμα των επικοινωνιών, η ε, προστασία του περιβάλλοντος, η άμυνα, η, ε, η ενέργεια, η προστασία της ειρήνης ασφαλώς στην περιοχή και η αξιοποίηση όλων των υφισταμένων μέσων για την περιοχή. Αυτό που μας αρέσει λιγότερο και ελπίζουμε να μπορέσουμε να διορθώσουμε είναι ότι δεν εμβαθύνουμε ιδιαίτερα στο θέμα που γίνεται όλο και πιο καυτό της παράτυπης, μετανάστευσης. Ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να ε, λάβει δική του θέση μέσα στην έκθεση και τη στρατηγική του κ. Ιάκοφτσιτς από την Επιτροπή της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ξέρετε ότι λύσεις σε αυτό δεν έχω να σας προσφέρω η Σύνοδος Κορυφής ασχολήθηκε με το θέμα της μετανάστευσης, αλλά και με τις ροές ε, και την ένταση της εγκληματικότητας. Θα ήθελα λοιπόν να ενσωματωθεί στο κείμενο το θέμα της παράτησης μετανάστευσης και της διασυνοριακής εγκληματικότητας, εκεί που γίνεται λόγος για τη στρατηγική, για τις, ε, στο κείμενο στρατηγικής για την περιφέρεια Αδριατικής Ιωνίου. Αυτό έχετε και τις ε, ε, τροπολογίες αν δεν απατώμε. Θα τις συστήσουμε ασφαλώς. Η Επιτροπή μας αναμένεται στις 15 Ιουλίου να συζητήσει και βεβαίως οτιδήποτε έχετε να συμπληρώσετε για την ε, συζήτηση με στη θέση σας. Ask Μη ζητάτε τροπολογίες, μπορεί να σας τις καταθέσουν. Παρακαλώ. Κύριε Σπιτσούλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Σουίτσα, για την παρουσίαση της γνωμοδότησής της. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω κιόλας για την διάσταση αυτή εξωτερικής πολιτικής ή τη γεωπολιτική που έχει συμπεριλάβει στη γνωμοδότησή της. Νομίζω είναι πλέον η τρίτη ε, μακροπεριφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καλύπτει μόνο τα οικονομικά ή θέματα μεταφορών, αλλά είναι εξόχως πολιτική. Τέσσερα κράτη-μέλη της Ένωσης καλύπτονται και γύρω στις 8 υποψήφιες χώρες, συνολικά 70 εκατομμύρια πολίτες. Και ακριβώς η συμμετοχή τους σε μια τέτοια ευρωπαϊκή διαδικασία είναι τόσο σημαντική γιατί φέρνει πιο κοντά την Ευρώπη. Ωστόσο, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και αντικειμενικές διαφορές μεταξύ των κρατών αυτών. Όχι μόνο ως προς την προθυμία τους ή την επιθυμία να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν και μακροοικονομικές διαφορές. Το δείχνουν άλλωστε και οι διάφοροι δείκτες ε, και κάθε χρόνο όλο και πιο σαφώς. Ε, εκτός αυτού, ορισμένα από τα κράτη αυτά στερούνται υποδομές ή εκεί που τις ε, διαθέτουν αυτές πολύ υπανάπτυκτες. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό από την ελόγω στρατηγική. Ε, ο αυτοκινητόδρομος Ατριατικής Ιωνίου είναι ένα σημαντικό έργο και ελπίζουμε να υποστηριχθεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν μπορεί έτσι στην τύχη να εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται την απαραίτητη υποδομή η ε, η περιφέρεια αυτή έχει φανεί ε, ότι είναι ευαίσθητη, φαίνεται και από τα stress test. Ε, επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία ο αγωγός φυσικού αερίου ε, Αδριατικής Ιωνίου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό το θέμα της ενέργειας. Εκτός από την ενέργεια αναφέρεται και το ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών. Οι μεταναστευτικές ροές νομίζω όμως θα πρέπει να διαχωριστούν από τις παράνομες. Βλέπουμε τις πρόσφατες εξελίξεις με την Ουγγαρία να υψώνει ένα τείχο στα σύνορά τη με τη Σερβία. Δεν μπορεί να είναι αυτή η λύση. Εγώ ποντάρω στο δυναμικό και στις δυνατότητες αυτές τη μακροοικονομική περιφέρειας και ελπίζω ε, να αντιμετωπιστεί και το θέμα της μετανάστευση. Ελπίζω όλοι οι ε, ενεχόμενοι να ενδιαφερθούν ε, για συνεργασία και αυτό θα ευνοήσει και την κοινωνική συνοχή και την οικονομική συνεργασία και την περιβαλλοντική αηφορία και βιωσιμότητα. Ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για τη σταθεροποίηση της περιοχής και την ανάπτυξή της. Ευχαριστώ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih u ime να Εγώ θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφο Σουίτσα για την έκθεσή της, αλλά και το κύριο Γιάκο Τσίση που είναι ο επί της ουσίας εισηγητής, εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για μια περιοχή ασταθή και ευάλωτη. Και υπάρχουν ανησυχίε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ανησυχούμε για όλες τις περιφέρειες, αλλά κυρίως για τούτη εδώ την περιοχή, πρόκειται για την Αδυτική και το Ιόνιο. Δεν χρειάζεται τώρα να επαναλάβω όσα είπε ο συνάδελφος Πίτσουλα σε σχέση με τις οδικές συνδέσεις σε αυτή την περιοχή. Αλλά θα ήθελα να τονίσω μια πτυχή που δεν ε, υπογραμμίστηκε αρκετά αφορά το γεγονός ότι η περιοχή αυτή μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ως διάβλος ενεργειακού ανεφοδιασμού. Η διασύνδεση λοιπόν αυτών των κρατών με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ σημαντική να την έχουμε υπόψη μας καθώς μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχουμε δηλαδή πηγές ενέργειας που περνούν από αυτή την περιφέρεια για να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ε, Εγώ θα συμφωνήσω συγχαίροντα την κυρία Σουίτσα για την εξαιρετική τη έκθεση και με του υπολείπου συναδέλφου που μίλησαν για την πολύ σημαντική πολιτική και στρατηγική θέση της ε, Δυτική θάλασσα και του Ιουνίου. Επίση, θα πρέπει να εργαστούμε προ τη μείωση των κοινωνικών διαφορών, τη βελτίωση τη συνοχή των Δυτικών Βαλκανίων, καθώ και πολλά άλλα στοιχεία που θα πρέπει κανεί να τονίσει. Όμως, θα ήθελα επίσης να αναφέρω την τροπολογία υπαριθμών 42 των πρασίνων καθώς αυτή αφορά την ποιότητα του περιβάλλοντος. Θέμα στο οποίο αυτή η περιοχή θα παίξει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ασφάλεια στην ενέργεια και τον ενεργειακό εφοδιασμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να στηρίξουμε την έρευνα για φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Αδριατική θάλασσα καθώς και να ε, εξετάσουμε πολλές άλλες πτυχές καλύτερης συνεργασίας, καθώς και να εργαστούμε περισσότερο για την μελέτη αντικτύπου, γιατί όλα αυτά θα επηρεάσουν και το περιβάλλον στην περιοχή και θα πρέπει να το προστατεύσουμε καλύτερα, να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα και γι' αυτό και χρειάζεται κοινό σχεδιασμός. Καλύτερη συνεργασία δηλαδή με το... την περιοχή αυτή για να μην ζημιωθεί αρνητικά, ζημιωθεί μάλλον η φύση. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που τα περιλάβατε όλα αυτά στην έκθεσή σας. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ως Ιταλός βεβαίως δεν μπορώ παρά να είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για αυτή τη στρατηγική που ξεκινά εκ νέου την ανάλυση για μια γεωγραφική ζώνη που μας είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Η συνεργασία με την άλλη όχθη της Αδριατικής είναι φυσικά για μας θεμελιώδη σημασία και γι' αυτό σας ευχαριστώ την εισηγήτρια της γνωμοδότησης αλλά και τον εισηγητή Γιάκοφ στην αρμόδια της Ουσίας Επιτροπή που το έχουν υπογραμμίσει. Και θέλω να υπογραμμίσω και κάτι που ήδη υπόθηκε εν μέρει από άλλους συναδέλφους και αφορά τις λήψεις της ε, ε, υποδομές. Ε, είναι καλό να μιλάμε για τις ελλείψεις στις οδικές μεταφορές αλλά και στις σειροδρομικές μεταφορές. Να θυμηθούμε τον διάδρομο Αδριατική Ιωνίου γιατί αυτός έχει αντίκτυπο όχι μόνο στην ε, κινητικότητα στην περιοχή αλλά και στον τουρισμό που θα μπορούσε κάλλιστα να αυξηθεί. Όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια δεν είμαι πάντοτε σύμφωνο 100% με τα όσα υπόθηκαν. Είναι αλήθεια ότι όσον αφορά τα χώρε που βρέχονται από την Δυτική και το Ιόνιο έχουν οικοσυστήματα ευάλωτα όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι ο όγκος εισαγωγών του τάπος δεν είναι τόσο ε, μεγάλος. Υπάρχει μάλιστα και μείωση της ζήτηση όσον αφορά το φυσικό αέριο. Και εξάλλου ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος είναι πολύ μεγάλος, γι' αυτό και είναι πολύ επικίνδυνο. Ε, δεν θεωρούμε λοιπόν ότι είναι θετική η, λύση αυτή, αν συγκρίνουμε με τους κινδύνους. Το ίδιο και όσον αφορά τους σταθμούς, τα δηληστήρια στην Αδριατική, που θα μπορούσαν να διαλύσουν την τουριστική βιομηχανία, γιατί πρόκειται για μια θάλασσα εξαιρετικά κλειστή και σε περίπτωση ατυχήματος θα χρειάζονταν δεκάδες χρόνια πριν να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το οικοσύστημα σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης ε, να μιλήσουμε σοβαρά και για το θέμα της ε, παράνομης μετανάστευσης, γιατί αυτός είναι ένας άξονας, ε, ένας διεύλος από τον οποίο μας αλλά και για τον Ισλαμικό εξτρεμισμό που δυστυχώς πλήττει κάποιες από τις χώρες της περιοχής και από αυτή την άποψη θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες αυτές. Είναι σημείο κλειδί για να μπορέσουμε να βρούμε κατάλληλη απάντηση και λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Σπλένκοβιτς. Ευχαριστώ και όλους ε, τους συναδέλφους. Ε, μια που μίλησαν όλοι οι Κροάτες συνάδελφοι που είναι παρόντες σήμερα εδώ, να μιλήσω και εγώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Γιάκοφσιτς και τους υπόλοιπους που εργάστηκαν σε αυτή την ε, προσπάθεια. Είναι αρμόδιος η στη Γίνεται λόγος για την Αδριατική και τον, το Ιόνιο. Εγώ από το 2000 παρακολουθώ αυτή τη στρατηγική μαζί με τον συνάδελφο Πίτσουλα και είδαμε τις πρώτες προσπάθειες που τελικά έγιναν στρατηγική και είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τη Βαλτική, ακολούθησε ο, Δύναβη, ο Δούναβης και τώρα είμαστε ε, στην Αδριατική και στο Ιόνιο. Θα πρέπει να δούμε ε, για μας ε, τι έχει σημασία. Κάτι που βλέπω για πρώτη φορά στη συνεργασία είναι ότι δίνεται έμφαση στη διαχείριση και στους μηχανισμούς διακυβέρνησης. Θα πρέπει αυτή να είναι σταθερή και μόνιμη. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε κάποιες χώρες να ε, εξελιχθούν περισσότερο. Έχω ε, ιδία εμπειρία ε, σε αυτά τα θέματα και νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις των χωρών που θέλουν να συμμετέχουν για να μπορούν να δραστηριοποιούνται περισσότερο. Εκτός αυτού ε, υπάρχει και το θέμα της πολιτικής διεύρυνσης. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Από τις χώρες αυτές τέσσερις είναι κράτη-μέλη ε, και τέσσερις είναι στη διαδικασία διεύρυνσης πιο προχωρημένη, λιγότερο προχωρημένη φάση. Και επίσης υπάρχουν και χώρες που ε, δεν συμμετέχουν άμεσα ε, στην προσπάθεια αυτή, όπως η Μακεδονία λέει ο κύριος Πλένκοβιτς ή το ε, Κόσοβο. δεν εντάσσονται απολύτως σε αυτή την προσπάθεια, αλλά θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποια δυνατότητα να ενταχθούν, γιατί δεν βρέχονται από τη ε, θάλασσα, ούτε η Σερβία άλλωστε, ε, αλλά η Σερβία στο παρελθόν ήταν, όπως ξέρετε, τμήμα της Ιουκοσλαβίας, όπως και το Μαυροβούνιο και καλό θα ήταν να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό από τη στρατηγική αυτή και θα ήταν κρίμα να εξαιρούνται κάποιες χώρες επειδή δεν βρέχονται από θάλασσα. και σε θέματα τουρισμού, μεταφορών κτλ. Ο Επίτροπος Χάν, όταν ήταν αρμόδιος στην περασμένη θητεία για την περιφερειακή ανάπτυξη, εργάστηκε ακριβώς σε αυτό το τομέα. Τώρα ε, είναι χατοφυλάκιο της κυρίας Κρέτσου. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό που μπορεί να αποτελέσει κλειδί για την ανάπτυξη της περιφέρειας ευρύτερα και να αποδειχθεί σταθεροποιητικός παράγων. Και για θέματα που έχουν να κάνουν με την παράτυπη μετανάστευση. Βέβαια εδώ αυτό το θέμα αφορά κυρίως την Ελλάδα και λιγότερο χώρες όπως την Κροατία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ και τους ηγητές. Και την εισηγήτρια. Η εισηγήτρια θέλει το λόγο. Κυρία Σακοράφα παρακαλώ. Συγγνώμη, σας ξέχασα. Η κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σουίτσα για την παρουσίαση της νομοδότησής της και να πω εξ αρχής ότι συμφωνώ σε αρκετά από αυτά που υπόθηκαν από τους συναδέλφους. Όμως θα ήθελα να πω και τούτο ότι είναι φανερό τόσο από το σχέδιο γνωμοδότησης όσο και από το πλήθος των τροπολογιών που ήδη έχουν κατατεθεί ότι δεν θέλει τη γνωμοδότηση αυτή να υποστήριξει πραγματικά τη λειτουργία της USER έτσι όπως έχει αποφασιστεί. Η επιδίωξη της προσθήκης νέου πυλώνα αυτού της μετανάστευσης στην θεματολογία της ε, USER, μια στρατηγική που μόλις τώρα ξεκινά τα πρώτα του βήματα και στάδια εφαρμογής, χωρίς να έχει εγκριθεί ακόμη ούτε ένα έργο μακροπεριφερειακού χαρακτήρα, θεωρώ ότι μόνο ζημιογόνος μπορεί να είναι για την ίδια τη στρατηγική και δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Πόσο μάλλον όταν η προσθήκη αυτή όσον αφορά στην ήδη αποτυχημένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική ε, έχει προδικάσει κάτι δική μου άποψη ότι η USER ε, θα αποτύχει εξαιτίας όλων αυτών. Επιπλέον μια τυχόν επέκταση της μακροπεριφέρειας απειλεί να αποπροσανατολίσει τη στρατηγική από τους σκοπούς της που όπως γνωρίζετε αποτελούν τον καρπό μιας δημόσιας διαβούλευσης αρκετά ευρείας. Γνωρίζετε πολύ καλά άλλωστε ότι για τους λόγους αυτούς οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Γιουσέρ και ο Επίτροπος κ. Χάν στη συνάντηση τον 2ο του 12 συμφώνησαν πως για να είναι επιτυχής η στρατηγική θα πρέπει στο αρχικό τουλάχιστον στάδιο να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα έργα μακροπεριφερειακού ενδιαφέροντος μέσα στους τέσσερις οριστέντες πυλώνες και μεταξύ των ιδρυτικών μελών της ΙΟΣΕ και μόνο. Ε, άλλωστε τα διδάγματα από τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές που ισχύουν και εννοώ της Βαλτικής θάλασσας και του Δούναβη δείχνουν ότι είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση σε έναν περιορισμένο αριθμό κοινών δράσεων και ευκαιριών και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής, η δέσμευση και ο ηγετικός ρόλος των χωρών που συμμετέχουν. Γιουσέρ, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για τις χώρες αυτές να προχωρήσουν στην διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασμού τους, αξιοποιώντας με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο τους πόρους της Ένωσης, τους εσωτερικούς πόρους της Ένωσης, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και αναπτύσσοντας τις εσωτερικές ενεργειακές υποδομές της, ιδίως τις πιο απομακρυσμένες και λιγότερο καλά συνδεδεμένες περιοχές της προκειμένου να πάυσει η οποιαδήποτε απομόνωση των συμμετεχόντων κρατών από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντα, θα ήθελα να τονίσω ότι κανένας δεν έχει αποκλείσει στο μέλλον την προσαρμογή της γιουσέης στις ανάγκες που θα παρουσιαστούν, ωστόσο εκτιμώ για τους λόγους που ανέφερα ότι στην συγκυρία την τωρινή μόνο ε, ζημιογόνο θα ήταν το οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο. Σας ευχαριστώ. Θέλει η συγκήτρια να απαντήσει, η συντάκτης. Ε, φυσικά. Και ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για όλα τα σχόλια. Με χαρά σημειώνω ότι άπαξ και μπορούμε να συνοηθούμε για τις ε, τροπολογίες θα αναλάβει και τις διαστάσεις και το, τη, τον όγκο που θα, ήθελε, που θα θέλαμε η εκθέση του κ. Γιακόψης γιατί μας ενδιαφέρει όλους αυτή η ζώνη, η Μεσόγειο στην οποία όλοι ζούμε. Θέλουμε να είναι η στρατηγική προς όφελος των πάντων και δεν θέλουμε να παραμείνει γράμμα νεκρό το σύνολο των προτασών μας. Ο κύριος ε, Πλένκοβιτς πολύ σωστά επισήμανε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί για μια σταθερή διακυβέρνηση και πρέπει με την θέση σε εφαρμογή της ε, στρατηγικής να αξιοποιήσουμε και την εμπειρία των επιτρόπων μα τη κυρία Κρέτσου και του κυρίου Χάν, ταυτόχρονα πρέπει να ενισχύσουμε τις υποδομές. Με καλές υποδομές νομίζω όλοι θα είμαστε κερδισμένοι. Και νομίζω ότι μπορούμε να μιλούμε για τον αυτοκινητόδρομο Αδριατικής Ιουνίου πάνω από όλα που αναφέρει και ο κύριος Πλένκοβιτς, γιατί είναι ένας διάδρομο ο οποίος ε, έχει συζητηθεί πολύ. Έχουν επενδύσει τα κράτη, κράτη-μέλη σε μεγάλο βαθμό πόρους δικούς τους Φερρυπίν για το οδικό δίκαιο, αλλά πρέπει, για δίκτυο, αλλά πρέπει και για το σιδηροδρομικό δίκτυο να αρχίσουν τα έργα. Και πρέπει να φτάσει το δίκτυο αυτό όλο, ο διάδρομος αυτός, μέχρι την Πάτρα, όπως υπόθηκε. Για το καλό της ειρήνης. Γιατί όλα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα αν υπάρχουν αυτές οι καλές υποδομές. Και αν ε, δημιουργηθούν πραγματικοί όροι συνοχή στην περιοχή. Βεβαίως τώρα έχουν ε, ακόμη πολλές ε, διαφορές μεταξύ τους στα κράτη αυτά. Πρέπει να κοιτάξουμε το κοσμοπέδιο και την ε, Μακεδονία, λέει ο Μιλήτρια, για να δούμε ποιος είναι ο ρόλος τους και πώς μπορούν να ενταχθούν στη στρατηγική. Και πρέπει να δούμε και τη Σερβία, που δεν έχει έξοδο ούτε στην Αδριατική, ούτε στην Μεσόγειο, ούτε στην στο Ιόνιο, αλλά είναι τμήμα των στρατηγικών αυτών. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά και είμαι βεβαία ότι θα υιοθετηθούν οι στρατηγικέ θα υιοθετηθεί η στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο, όταν μπορέσουν και οι λοιπέ επιτροπέ να ολοκληρώσουν την εκπόνηση των κειμένων του. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσαμε και αυτό το θέμα της ημερήσια διάταξης. Βλέπω να τελειώνουμε πιο γρήγορα από ό,τι πρόβλεπα. 15 Ιουλίου προθεσμία. Μάλλον ψηφοφορίες η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει να ψηφίσει 19 Σεπτεμβρίου και άρα υπάρχει αρκετό χρόνο, όπω βλέπετε, αγαπητοί συνάδελφοι, για την κατάθεση των τροπολογιών. Έχουμε τελειώσει τώρα για τι συζητήσει μα. Οι ψηφοφορίε που βλέπονται για τι 6 το βράδυ, δυστυχώ θα πρέπει να διακόψουμε, αφού φαντάζομαι ότι θα έχουν οι συνάδελφοι προβλέψει να έρθουν στι 6 για την ψηφοφορία. Δεν μπορώ να ξεκινήσω νωρίτερα τι ψηφοφορίε, πιστεύω να συμφωνείτε κι εσεί.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 ποτέ δεν Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Κυρίες και κύριοι. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε. Thank you for coming back. Σας ευχαριστώ που επιστρέψατε. Έχουμε την τελική ψηφοφορία για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου 1236 κάθετος 2005 για το εμπόριο ορισμένων αγαθών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Και όποιος έχει καταλάβει αυτό τον τίτλο έχει και το προνόμιο να ψηφίσει. κυρία Λόχμπίλερ, θέλετε να πείτε τίποτα? Ευχαριστώ όλους κοιόδης ήταν πάρα πολύ καλή η συζήτηση και σήμερα η Ίντα που είναι επί της ουσίας αρμόδια το συζήτησε για πρώτη φορά και έχουμε συναντήληψη πάνω κάτω για τα περισσότερα θέματα. Α, Ίντα είναι η Επιτροπή και αυτό δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα, αλλά ας ψηφίσουμε τώρα. Yeah. Ο κύριος Κόρβεν Μίκε. Μα οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν νερό για να βασανίζουν τους κρατουμένους. Το νερό δεν το έχει αυτός ο κατάλογος εδώ πέρα. Ε, το waterboarding το περίφημο. <laughs> So, let's vote. Υπάρχει και το vodka board. Λοιπόν, ψηφίζουμε 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 και 38 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 και 39 είναι οι ίδιες και αυτές. Έλεγχο θέλετε για τις δύο προηγούμενες. Die Abstimmung ist geschlossen. ψηφοφορίας. you your credit card again? Πάλι την πιστοτική σου έβαλες, Γιάτσακ. we have to start again. Something... Αρχίζουμε, γιατί κάτι πήγε στραβά, ξανά. Πάλι όλοι παρακαλώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Τώρα τελείωσε. Έγκρινεται 28 υπέρ 17 κατά. Τροπολογία 3 και 39 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 και 10 λέει ο πρόεδρος. Όχι, 4 και 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 42 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Ευχαριστώ, κατά Αποχές συγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο θέλετε καλώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 24 υπέρ 25 κατά. Και ήταν αυτή η 42. Πάμε στη 5. Ψηφίτε. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Την 5 παρακαλώ. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. Es wird 29 zu 19 angenommen. Εγκρίνεται 29-19. Η 6 είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 και 43 μαζί είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 46 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 και 48 είπε. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 24 υπέρ, 21 ε, κατά. Η συμβαστική 1 Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 10 μαζί με την 51. Ψήφιπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 55 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Die Abstimmung ist geschlossen. Απορρίπτεται 23 υπέρ, 27 κατά. Η 56 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Η 11 και 58 μαζί υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η τροπολογία 60 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 61 είπε. Υπέρ 61. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 61 παρακαλώ. Die Abstimmung ist geschlossen. 23, 26 Απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά, κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Α, σωστά. Συμβιβαστική 2 πρώτα. την έχασαμε στον γκρι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 72 υπέρ, κατά, αποχές, Απερίφθη 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαληθεύουμε τη συμβαστική 4. 29 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά. Α, με συγχωρείτε, συμβαστική 5. Αυτό το γκρι δεν το βλέπω ποτέ. Να βάλω καλύτερα γυαλιά. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 23 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 26 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 27 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 28 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 29 υπέρ κατά αποχές. Ε, επαληθεύουμε. Πέρας. Απεριφθεί. 24 ψηφί, υπέρ, 25 κατά. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Πέρας. 23 υπέρ. 27 κατά απερίφθη. 33 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Και ηλεκτρονικά την τελική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 45 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, 3 εποχές. Εγκρίνεται και ευχαριστούμε πολύ την συγκεντρία. Προσεχή συνεδρίαση στις 15 Ιουλίου, πέρα στη συνεδρία σας.